Είναι 12 λεπτά πριν τις 5. Σας καλωσορίζω όλους μπροστά στις οθόνες των υπολογιστών σας. Ερχόμαστε στην ανακοίνωση του αποτέλεσματος της πρώτης ψηφοφορίας για σήμερα το πρωί. Εγκρίθηκαν εξής τροπολογίες και οι δύο όλες μάλλον από την 1 μέχρι την 41 μετά και οι τροπολογίες 10, 11, 103, 191, 226, 227, το πρώτο μέρος. Οι εξή τροπολογίες απερίφθησαν. 188. 4, 188, 35, 59, 65, 95, 98, 104, 106, 124, 135, 144, 158, 192, 227, το δεύτερο μέρος. Ένα τμήμα 41, 248 ε, καταπίπτει επειδή ε, εγκρίθηκε στη συμβιβαστική 41 το αντίστοιχο μέρος. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της πρωινής ψηφοφορίας από πλευράς μου. Προχωρούμε ε, στη δεύτερη ψηφοφορία τώρα που θα αρχίσει από τις 5 μέχρι τις 6.30 θα διαρκέσει. Ξέρετε τη διαδικασία με το ψηφοδέλτιο. Το αποτέλεσμα της ε, τελικής ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί γραπτός. Ξέρετε πώς στέλνετε ε, το ψηφοδέλτιο από την επίσημη διεύθυνσή σας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο γνωστό ε, σημείο. Μέχρι τις 6.30, από τη στιγμή που θα ανοίξει η ψηφοφορία στις 5. Αυτή τη στιγμή, αν ανοίξει η ψηφοφορία, θα λάβετε mail που θα επιβεβαιώνει ακριβώς την έναρξη της ψηφοφορίας. Οι παρόντες, που δεν υπάρχει κανένας εκτός από μένα, ε, πρέπει να ψηφίσουν και αυτοί γραπτός και θα σας ανακοινθούν ε, τα αποτελέσματα. Για να διαπιστώσουμε παρακαλώ την απαρτία που είναι 18 μέλη. Σας παρακαλώ ε, πατήστε το κουμπί που λέει ζητώ το λόγο το χεράκι για να δούμε αν έχουμε απαρτία τώρα. Άλλον έναν, σας παρακαλώ, χρειαζόμαστε για την απαρτία. Excellent. We are done. Εξαιρετικά. Διαπιστώνεται η απαρτία. Διαπιστώθηκε και εξακριβώθηκε η απαρτία. Αρχίζει ψηφοφορία και έχετε χρόνο μέχρι τις 6.30 για να ε, στείλετε τα ψηφοδέλτιά σας. Ο Επίτροπος είναι έτοιμος. Ο Επίτροπος Βάρχελη έχει συνδεθεί. Mr. Commissioner, could you please press the hmm? Yes. Επίτροπος, παρακαλώ. Επίτροπε, αγαπητέ Όλιβερ, με χαρά σας καλωσορίζω και πάλι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στο διάλογο για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Θέλουμε να συζητήσουμε την κατάσταση στο Μαυροβούνιο πρώτα και μετά στη Σερβία. Έχετε γνώση ε, του γεγονότος ότι και εμάς μας ενδιαφέρουν πολύ τα Δυτικά Βαλκάνια όπως και σας, και το Μαυροβούνιο. Πριν την πανδημία είχαμε προγραμματίσει το Μάιο αποστολή στην Ποτγκόριτσα που δυστυχώς ματαιώθηκε. Αλλά το Μαυροβούνι παραμένει ψηλά στη δική μας ε, ημερήσια διάταξη και στα ενδιαφέροντά μας. Στις 30 Αυγούστου είχαν βουλευτικές εκλογές με μεγάλη συμμετοχή παρά την πανδημία και τις απαιτητικέ ε, συνθήκες. Πριν τις εκλογές είδαμε πολύ πολλωμένο το κλίμα και συζήτηση για την παράθεση για θέματα εκκλησίας και εθνικής ταυτότητας. Μετά τις εκλογές που έδωσαν πλειοψηφία σε μια, ένα συνασπισμό της αντιπολίτευσης, βλέπουμε κόμματα, τώρα πώς να το πω, που έχουν εξαιρετικά διστάμενες πολιτικές απόψεις αυτό κάπως ε, θορύβησε τις Βρυξέλλες. Καλωσορίζω το γεγονός ότι ο νέος ε, κυβερνητικός συνασπισμός ε, υπέγραψε μια συμφωνία. Συμφωνούν τα κόμματα να παραμείνουν προσιλωμένα στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Τις επόμενες εβδομάδες θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή η κυβέρνηση, νομίζω στις 2 Δεκάτου και ελπίζουμε να είναι μεγάλη και διακομματική η συμφωνία για τις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από το πακέτο της διεύρυνσης κάνουμε και έκθεση ε, για το Μαυροβούνιο για το 2019 και 2020. Γι' αυτό η σημερινή συζήτησή μας είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Ε, οι συνάδελφοι επίσης ενδιαφέρονται πολύ να μας πείτε τι έγινε στη Σόφια ε, στη Σύνοδο Κορυφής της 10 Νοεμβρίου για τη διαδικασία του Βερολίνου, ε, ε, τα Δυτικά Βαλκάνια, την Πράσινη Ατζέντα και την Κοινή Περιφερειακή Αγορά. Θα σας δώσω το λόγο τώρα για 10 λεπτά και στη συνέχεια στους συναδέλφους που έχουμε στον κατάλογο ψηφοφορίας και θα απαντήσει ο Επίτροπος στις ερωτήσεις μας. Χρόνο έχουμε για το Μαυροβούνιο μέχρι τι 6 παρατέταρτο, 50 λεπτά δηλαδή, και από τις 6 παρατέταρτο μέχρι τις 6.30 έχουμε αντίστοιχη συζήτηση για την κατάσταση στη Σερβία. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, που ήρθατε στην Επιτροπή μας ε, διαδικτυακά. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, David. Ε, και ελπίζω να είναι η μοναδική φορά που να μιλάμε εξ αποστάσεω. Την επόμενη φορά ελπίζω να μπορέσω να είμαι παρόν για να συζητήσουμε τα θέματα κοινού ενδιαφέροντο. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και πάλι στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Σας ευχαριστώ και πάλι που συνεχίζετε να εργάζεστε ε, με συνέπεια παρότι ε, πρέπει να προσαρμοστείτε στις ε, συνθήκες. Να αναφερθώ λίγο στα Δυτικά Βαλκάνια προτού φτάσω στο σημερινό θέμα, την κατάσταση στο Μαυροβούνιο και κατόπιν στη Σερβία. Πριν από ένα μήνα σας παρουσίασα το οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια μέχρι 9 δισεκατομμύρια ε, παρήχαμε, τα οποία ε, θα συμπληρωθούν από την ε, νέα διευκόλυνση εγγύησης για τα Δυτικά Βαλκάνια που θα πρέπει να μπορεί να συγκεντρώσει επενδύσεις μέχρι 20 δισεκατομμύρια. Η μόχλευση Ε, αυτών των επενδύσεων ε, θα πρέπει να μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ της περιοχής ε, κατά 3,6%. Μια κοινή περιφερειακή αγορά είναι ο στόχος που να ενσωματώνει και την πρωτοβουλία Mini Schengen καθώς και πράσινο θεματολόγιο για τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάνω στα δύο αυτά θέματα ήδη βλέπουμε θετική ανταπόκριση και Επίση, ε, πολιτική δέσμευση. Την προηγούμενη εβδομάδα, στη διάσκεψη κορυφής της ε, Σόφιας, ε, συμφωνήθηκε ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την κοινή περιφερειακή αγορά, για ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, υπηρεσιών, ανθρώπων και κεφαλαίων. Θα αυξήσει την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα των Δυτικών Βαλκανίων θα γίνουν κόμβος επενδύσεων ε, που θα προσελκύουν ε, διεθνείς επενδυτές. Οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων επίσης ε, υιοθέτησαν το πράσινο θεματολόγιο καθώς και προτάσεις για ψηφιακή μετάβαση για την νεολαία, την καινοτομία, την επιστήμη και με το πράσινο θεματολόγιο δεσμεύτηκαν να ε, ε, στοχεύσουν στο δικό μας ε, στόχο για το κλίμα, δηλαδή κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Ε, επίσης, όσον αφορά τους Ρωμά, στα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχουν οι περισσότερες οικογένειες Ρωμά χωρίς δουλειά εδώ και γενιές αλλά για να έχουν πραγματικές ευκαιρίες ε, στην κοινωνία ε, υπάρχει τεράστιο περιθώριο ε, βελτίωση και θα πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτό το σχέδιο. Το οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν την περιφέρεια οδηγώντας σε μια πιο ψηφιακή και πιο ζωντανή οικονομία. Επιπλέον λαμβάνουμε κάποια πρώτα βήματα προς ε, την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου με το ε, σχέδιο συνδεσιμότητας 2020 που περιλαμβάνει έξι προγράμματα για βιώσιμες ε, μεταφορές και πράσινη ενέργεια. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει η επενδυτική αυτή δέσμη. Να μιλήσω τώρα για το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο έχει ξεκινήσει και τα 33 κεφάλαια και προσωρινά έχουν κλείσει τρία από αυτά. Στην μετεκλογική περίοδο η νέα κυβέρνηση και το νέο κοινοβούλιο πρέπει να ε, πετύχουν ε, ε, διακομματική και ευρέως αποδεκτή συνένεση για την εφαρμογή του θεματολογίου. Να ξεκινήσω από το, την οικονομική κρίση που οφείλεται στην πανδημία του κορονοϊού. Είναι πολύ δύσκολες οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, ε, καθώς ε, και οι προσπάθειές μας για να βοηθήσουμε το Μαυροβούνιο. 20% του ΑΕΠ έχει χάσει η χώρα λόγω της ε, κρίσης του κορονοϊού. Λόγω του ε, κυρίαρχου ρόλου του τουρισμού στην οικονομία επιπλέον, το χρέος της χώρας ε, γίνεται όλο και πιο ανησυχητικό. Θέλουμε να παράσχουμε επίγουσα βοήθεια στο Μαυροβούνιο και δεύτερον, να ε, ανακάμψει η οικονομία. Το πρώτο κύμα υποστήριξης από εμά είχε στόχο την παροχή επίγουσας γιατρικής βοήθειας, ενώ το δεύτερο κύμα ε, στόχο είχε να βοηθήσουμε το Μαυροβούνιο να ξεπεράσει τις άμεσες ε, συνέπειες ε, του κορονοϊού λόγω της εξάρτησής του από τον τουρισμό. Ως τμήμα της βοήθειας αυτής για οικονομική ανάκαμψη, την προηγούμενη εβδομάδα στις 10 Νοεμβρίου δώσαμε 28 εκατομμύρια και 53 εκατομμύρια έχουν δοθεί συνολικά σε επιχορηγήσεις και 60 εκατομμύρια σε μακροοικονομική βοήθεια. Να αναφερθώ τώρα στο πολιτικό περιβάλλον στο Μαυροβούνιο και τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Το Μαυροβούνιο μετά τις εκλογές της 30 ε, ε, Αυγούστου βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο. Ε, ήταν πολύ μεγάλη η προσέλευση των ψηφοφόρων, 76% ε, αποτελεί ρεκόρ αυτό. Οι διεθνείς παρατηρητές επεσήμαναν ότι υπήρχε διαφάνεια στις εκλογές. Το αποτέλεσμα των εκλογών ε, ήταν μια αναπάντεχη αλλαγή όσον αφορά την κυβερνητική συμμαχία. Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της νέας χώρας υπάρχουν διάφορες ε, λύσεις ε, για το σχηματισμό κυβέρνησης. Ο κύριος Μπέτσιτς είναι νέος πρόεδρος του Κοινοβουλίου και αυτό είναι ένα βήμα που επικροτούμε όσον αφορά τους ε, θεσμούς. Ο καθηγητής Κλεβοκάπιτς ε, ε, έχει οριστεί πρωθυπουργός. και έχει προσπαθήσει να συγκεντρώσει το σύνολο τη ε, πρώην αντιπολίτευση για να σχηματίσει κυβέρνηση. Οι προσπάθειέ του για σχηματισμό κυβέρνηση συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να επικροτήσω το γεγονό ότι ο συνασπισμό των πρώην κομμάτων της αντιπολίτευσης ε, υπέγραψε δημόσια διακήρυξη όπου δεσμεύονται να τηρήσουν τις ε, διεθνείς υποχρεώσεις ε, του Μαυροβινίου, ιδιαίτερα όσον αφορά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι θετικό σημάδι, διότι υπάρχει διακομματική υποστήριξη και γενική υποστήριξη από την κοινωνία στο σύνολό της. Αναμένουμε λοιπόν μεταρρυθμίσεις οι οποίες απαιτούν ε, ειδική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Προσβλέπω και στην πλήρη ευθυγράμμιση του Μαυροβουνίου με την ε, ευρωπαϊκή πολιτική, το οποίο ήδη έχει αποτελέσει πολύ ε, σημαντικό μήνυμα από πλευρά τη χώρα. Αρχέ του Νοεμβρίου, ο διοριστή Πρωθυπουργό έχει ε, ανακοινώσει ότι 12 υπουργού θα έχει κυβέρνηση. Πολλοί από αυτού ε, είναι νέοι άνθρωποι και θα πρέπει κατά την κοινοβουλευτική σύνοδο στις 2 Δεκεμβρίου να ε, συζητηθούν τα θέματα αυτά. Όποια και αν είναι η σύνθεση της νέας κυβέρνησης θα αντιμετωπίσει δύο βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη είναι η εμβάθυνση και η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα στο, ε, στον τομέα του κράτους ε, δικαίου και Ιδιαίτερα μα ενδιαφέρουν εδώ πέρα τα σημεία αναφοράς για τα ε, κεφάλαια 23 και 24 και το δεύτερο είναι ε, το να ξεπεραστεί η κοινωνικο-οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού που έχει ε, χτυπήσει πολύ βαριά το Μαυροβούνιο. Αυτές οι προκλήσεις απαιτούν μια δημόσια δομή η οποία να λειτουργεί καλά και ε, χρειαζόμαστε μια γρήγορη μετάβαση, ένα μήνυμα το οποίο συνεχώς μεταφέρω στους ε, πολιτικούς ηγέτες στην Ποτκόριτσα εδώ και μήνες η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μαυροβούνιο. Ε, καλεί την νέα κυβέρνηση να ξεκινήσει γρήγορε εργασίες της και περιλαμβάνει και προτάσεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να κινηθεί. Προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία με το νέο Κοινοβούλιο και τη νέα κυβέρνηση για να προχωρήσουν γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την προσχώρηση. Συνεχίζουμε να είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι όσον αφορά να είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι όσον αφορά την διαδικασία προσχώρησης ε, του Μαυροβουνίου ε, καθώς ε, και να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να ανακάμψει από την κρίση. Θα κλείσω εδώ προς το παρόν, θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε, Όλιβερ Βαχέλη, τον Επίτροπο για τα εισαγωγικά του σχόλια μετά τις εκλογές. Στο Μαυροβούνιο έχουμε τώρα χρόνο για ανταλλαγή απόψεων και μετά, ε, θυμίζω από το σημείο αυτό, θα συζητήσουμε τη Σερβία. Τώρα θα δώσω το λόγο στους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών, των επαγγέλευση της αντιπροσωπίας μάλλον για τις σχέσεις με, τον, με το Μαυροβούνιο, τον κύριο Μπίλσεκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Ντέιβιντ, ελπίζω να με ακούτε και να με βλέπετε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι πολύ καλή αυτή η ευκαιρία να έχουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή ανταλλαγή για την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι σημαντικό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και πρέπει να δείχνουμε και τη στήριξή μας για τους εταίρους μας στην περιοχή αυτή και για το Μαυροβούνιο που υπήρξε για πολλά χρόνια, ηγείτο μάλλον για πολλά χρόνια της διαδικασίας ε, αλλά επλήγει προσχώρησης, αλλά επλήγει ιδιαίτερα από την ε, κρίση της ε, πανδημίας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προκειμένου η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας να είναι να παραμείνει ζωντανή, να παραμείνει στην τροχιά της. Τώρα, Λυπάμαι φυσικά που τα μέλη του Κοινοβουλίου δεν μπορούσαν να είναι στο Μαυροβούνιο τον Αύγουστο για να παρακολουθήσουν τις εκλογές λόγω της πανδημίας. Αλλά εκφράζουν ικανοποίησή μου ότι είχαμε πολύ καλά διοργανωμένες εκλογές στο Μαυροβούνιο. Οι πολίτες ε, προσήλθαν σε ποσοστά ρεκόρ η συμμετοχή τους ήταν πάρα πολύ υψηλή και τελικώς υπερψήφισαν την πολιτική αλλαγή. Ήταν πολύ μεγάλα τα νέα αυτά για τη χώρα αλλά και συνολικά για την Ευρώπη. Και αυτά τα μεγάλα νέα είναι και καλά νέα πιστεύω για το μέλλον του Μαυροβουνίου και είναι μια ευκαιρία να θέσουμε τα σχόλια μας, παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις μας ιδιαίτερα προς τον Επίτροπο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και οι πολίτες της. Καταρχά, πολύ χαίρομαι που ξεκινήσατε με την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση. Και η ερώτησή μου είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να κινητοποιήσουμε και τους διεθνείς φορείς, τους οικονομικούς, ώστε το Μαυροβούνιο να λάβει την βοήθεια που χρειάζεται, προκειμένου να επιβιώσει γιατί το διακύβευμα την κρίση αυτή είναι το πολιτικό μέλλον της χώρας στην ουσία. Με τις φιλοδυτικές, φιλοευρωπαϊκές τάσεις που έχει και τις οποίες πρέπει να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε χωρίς να καθυστερήσουμε γιατί εδώ υπάρχει μια ευκαιρία και για εξωτερικές δυνάμεις να παρέμβουν στο παιχνίδι. Επομένως η Επιτροπή τι σχεδιάζει να κάνει ως προς αυτό. Ως προς το COVID και όχι μόνο συγκεκριμένα για το Μαυροβούνιο, πώς είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε και τους δικούς μας πόρους και μέσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, ιδιαίτερα όταν θα έχουμε ένα εμβόλιο. Δηλαδή έχουμε ένα σχέδιο για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς με τα μέσα που, έχουμε, που θα έχουμε στη διάθεσή μας για να βοηθήσουμε το Μαυροβούνιο και άλλες χώρες περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος τον κύριο Μπίλτσεκ θα ακούσουμε και πάλι, θα τον ακούσουμε και πάλι στο επόμενο σημείο και πάω στον πρώτο γύρο των συντονιστών ή των συναδέλφων που τους αντικαθιστούν ο κύριος Ντέλη. Καταρχάς για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ αγαπητέ Ντέιβιντ, αγαπητέ Επίτροπε. Συνάδελφοι, ως προς το Μαυροβούνιο, δεν μπορεί κανείς να υπογραμμίσει αρκετά ότι πρόκειται για μία από τις χώρες που ηγείτο στη διαδικασία της διεύρυνσης. Και το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατάφεραν να σημειωθεί πρόοδος και να έχουμε ανοίξει κεφάλαια. Χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και οικονομική ενίσχυση. Ως προς την πολιτική σταθερότητα περιμένω με ενδιαφέρον να δω τη νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί 2 Δεκεμβρίου και ελπίζω να έχουμε σταθερότητα μετά από αυτό. Το ΕΛΚ και το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να, έτοιμα να βοηθήσουν τους φίλους μας ε, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά στο Κοινοβούλιο της Ποντγκορίτσα. Τώρα, οικονομικός μιλώντας, η κατάρρευση του ΑΕΠ, ε, ιδιαίτερα λόγω φυσικά της κατάρρευσης της τουριστικής βιομηχανίας, ήταν πολύ σημαντική. Πρέπει να ενισχύσουμε το Μαυροβούνιο και αυτό είναι προφανές, αλλά τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε, αυτή είναι η ερώτησή μου. Δηλαδή, το σημερινό πλαίσιο παροχής οικονομικής βοήθειας, πώς μπορούμε να το διευρύνουμε, γιατί ρεαλιστικώς μιλώντας είναι μια σημαντική χώρα αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη. Άρα το πρόσθετο άχθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν... δεν θα ήταν υπερβολικό. Και ήθελα να ακούσω τη γνώμη του Επιτρόπου επ' αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Άντορ. Για το S&D, ο κύριος Σίντα για δύο λεπτά. Κύριε Σίντερ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ναι. Ε, το πατούσα, αλλά δεν άνοιγε ε, το μικρόφωνο. Τώρα λειτουργεί. Αγαπητέ Επίτροπε, στα αγγλικά ο κύριος Σίντερ, αξιότιμε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε τις εκλογές στο Μαυροβούνιο και διαπιστώσαμε ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ πολλωμένο το κλίμα. Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας ήταν πολύ μεγάλος, πρωταγωνιστικός και είδαμε και εθνικιστικά επιχειρήματα να κυριαρχούν κατά τις εκλογές. Αυτή την τάση τη διαπιστώνουμε και σε άλλες γειτονικές χώρες, ε, αλλά και πιο πέρα όπως είναι η Βουλγαρία και λοιπά στα Βαλκάνια. Εμείς τι περιμένουμε. Τώρα τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, την οποία θα δούμε. Μπορεί να έχουμε λιγότερες μειονότητες να εκπροσωπούνται ε, σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο εθνικισμός, όπως γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο δηλητήριο για την περιοχή, ειδικά για το Μαυροβούνιο. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η στρατηγική ε, και στις προνταξιακές ε, διαπραγματεύσεις για να αποκρούσουμε τις ε, εθνικιστικές κορώνες. Και στη συνέχεια γνωρίζουμε ότι το Μαυροβούνιο έχει ανοίξει βέβαια όλα τα κεφάλαια, αλλά δεν τα έχει κλείσει. Τρία μόνο. Έχουμε πόρο από το να κλείσουν όλα τα κεφάλαια. Και τίθενται και, εκεί ερωτήματα τι μπορούμε να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τη νέα κυβέρνηση, όπως και στα άλλα θέματα, να επιταχύνει και τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Το σημαντικό δεν είναι να ανοίγουν τα κεφάλαια, αλλά να κλείνουν και να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Thank you. Ευχαριστώ, Ανδρέα Σίντερ, για τα σχόλιά σας. Από την ομάδα Renew, ο Ιλχάν Κιουτσουκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους συνάδελφοι και σας Επίτροπε και ευχαριστώ που βρήκατε το χρόνο για μας. Είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Πάντα είναι επίκαιρη συζήτηση για τα Δυτικά Βαλκάνια. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που λένε ότι είναι δύσκολη καιρή μπροστά μας κιόλα για την πανδημία COVID αλλά και τα οικονομικά προβλήματα ε, του Μαυροβουνίου και των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και οι συνθήκες πανδημίας ε, άσκησαν το δημοκρατικό τους δικαίωμα οι πολίτες και ψήφισαν νέα κυβέρνηση, ε, νέο κοινοβούλιο δηλαδή πρώτα και θα αναλάβει νέα κυβέρνηση. Έγινε ε, ένα πρώτο βήμα με το κυβερνητικό συνασπισμό. Έχει προχωρήσει πολύ στην ενταξιακή διαδικασία το Μαυροβούνιο και για μας είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια θα είναι η νέα κυβέρνηση και θέλουμε να επιταχύνει τις οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα έπεσε πολύ λόγω COVID ε, η οικονομία, τα έσοδα. Εσείς τι περιμένετε τώρα με αυτή την αλλαγή της κυβέρνησης. Θα επιταχύνει την ενταξιακή της ε, πορεία της χώρας ή όχι. Και πώς βλέπετε τη σχέση Σερβίας-Μαυροβουνίου. Είχαμε σκαμπανεβάσματα σε αυτή τη σχέση. υπάρχουν τριβές στι σχέσεις με τη Σερβία. Συγγνώμη που θα τα πω ομά, επίτροπε. Αυτό το ενδεχόμενο βέτο ή το βέτο της Βουλγαρίας για τη Βόρεια Μακεδονία θα επηρεάσει χώρες όπως το Μαυροβούνιο που θεωρείται ε, ότι πρωτοστατεί και είναι κοντά, ε, έχει προχωρήσει στις προενταξιακές. Ε, η κυρία Μπίλτ από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας είχα κάνει μια γραπτή ερώτηση για το σχέδιο αυτοκινητοδρόμου 800 εκατομμύρια ε, ευρώ κοστίζει και έχει ολέθριες συνέπειες για τα οικονομικά της χώρας. Φτάνει περίπου το 100% του προϋπολογισμού της χώρας, ε, με του ΟΕΠ, ε, για το 2021 και μάθαμε ότι και εκεί να ενδιαφέρεται για το κεντρικό θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο. Κάτι αντίστοιχο ε, μας θυμίζει και στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Πώς θα μειωθούν έτσι οι εκπομπές. Βάζει χέρι όλο και περισσότερο στο Μαυροβόνιο η Κίνα. Αυτό δεν αντιτίθεται με μια ενδεχόμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και η παγίδα του χρέους, είναι κίνδυνος. Τι γίνονται με τα μεγάλα έργα ε, και ιδιαίτερα τα θερμοελεκτρικά που βασίζονται στον άνθρακα και προωθεί η Κίνα στα Βαλκάνια. Ανησυχούμε ε, για την υποχώρηση των δημοσίων ελευθεριών λόγω πανδημίας. Το έχετε συζητήσει αυτό με τις αρχές της χώρας. Έχουν συλλάβει ιερείς ε, ορθόδοξους επειδή έκαναν λειτουργία. Αυτά είναι υπερβολικά και δείχνουν και μια διαλαξία απέναντι στην Εκκλησία μετά από τον πάρα πολύ αμφιλεγόμενο νόμο για τις εκκλησίες ε, που πέρασε το Μαυροβούνιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τόμας Βάιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ξαναήρθατε στην Επιτροπή μας. Έχω κάποιες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις να θέσω. Ο οριστής Πρωθυπουργό είναι πολύ δραστήριος, προσπαθεί να σχηματίσει η κυβέρνηση. Είχατε συνομιλίες μαζί του. Σημερίζεστε τη θέση ότι ε, στα σοβαρά σκοπεύει να ε, ε, επιδιώξει προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, στο ΝΑΤΟ. Θα ήθελα πολύ την προσωπική σας εκτίμηση. Πώς βλέπετε τις προσπάθειές του σε σχέση με κάποια κόμματα της μειοψηφίας που δεν θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση. αλλά επίσης ε, ο αντιπρόεδρος που σκοπεύει να ορίσει που θα είναι ε, αρμόδιος και για θέματα άμυνας θεωρείται ότι αυτό είναι θετικό βήμα απέναντι στις ε, μειονότητες και... Κάποιες θέσεις ανάλογες με τους υφυπουργούς σε άλλες χώρες. Μία θέση υφυπουργού για ανθρώπινα δικαιώματα και μία για ε, διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, θέματα, είναι αρμοδιότητες που θα ε, αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά θα υπάρχει και ένας υφυπουργό στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ε, βλέπετε, θεωρείτε ότι αυτά είναι σωστά βήματα για τη συμπερίληψη των μειονοτήτων και όσον αφορά τον ε, τομέα της ασφάλειας Ε, υπάρχει ένα κόμμα ιδιαίτερα φιλοευρωπαϊκό που φαίνεται ότι θα αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας. Ε, πιστεύετε ότι έτσι θα υπάρχει φιλοευρωπαϊκή θέση απέναντι και στο ΝΑΤΟ που δεν με ενδιαφέρει τόσο ε, ε, προσωπικά, αλλά και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς βλέπετε την συνεργασία στον τομέα της ασφαλείας και τελευταία ερώτηση. Ένας ε, υποψήφιος Υπουργός Εσωτερικών ε, ήδη αποσύρθηκε. Ε, τρόμαξε με το έργο που τον περιμένει, διότι σημαίνει ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα και την διαφθορά σε υψηλό επίπεδο. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε έναν Υπουργό Εσωτερικών για να μπορέσει να, το να επιτελέσει το έργο του. Και τέλος, ο Μάρκοβιτς και ο Γιουκάνοβιτς φαίνεται να ακολουθούν με πολύ δίκαιο τρόπο την ε, νέα ε, πλειοψηφία. Σημερίζεστε τη θέση αυτή. ότι παίζουν πολύ σωστά το δημοκρατικό της ρόλο σε αυτές τις νέες διαπραγματεύσεις ε, για κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τόμας Βάιτς. Χέρμαν Τέρτς από το ECR, παρακαλώ. I Με ενημερώνουν ότι δεν είναι συνδεδεμένος ο κύριος Τέρτς Από την ΓΚΟΕ δεν έχουμε ομιλητή, αλλά από τους μη εγγεγραμμένους μπορώ να δώσω το λόγο στον Φάμπιο Καστάλτο. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Βαρχέλη. Είναι κρίσιμη στιγμή, όπως επισημάνατε, για το Μαυροβούνιο, διότι με τις εκλογές αυτές έχουμε ε, μεταβάσει της εξουσίας ε, στην χώρα. Ε, είχαμε μια αποστολή παρατήρησης ε, παρακολούθησης ε, των εκλογών και εγώ παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις στη χώρα είναι σαφές ε, ότι για τον ε, συνασπισμό που κέρδισε τις εκλογές ε, τα δύσκολα τώρα ξεκινάνε. θα πρέπει να ασχοληθεί με τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, ο Τράφο Πιβοκάπιτς, ο Οριστή οριστής πρέπει να σχηματίσει η κυβέρνηση με υπουργού που να γίνουν αποδεκτοί από τους συμμάχου του. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε περισσότερε πληροφορίε σχετικά με τι διαπραγματεύσει αυτέ. Ε, όπως ε, αναφέρθηκε νωρίτερα, ε, τα κόμματα εθνοτικών μειοψηφιών αρνούνται να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση για πρώτη φορά από το 1998. Έτσι γίνονται κάποιες ανησυχίες σχετικά με πιθανό εθνικισμό. Αν ε, δεν εκπροσωπούνται αυτές οι μειονότητες θα αποκλειστούν τελείως ε, από τη δημοκρατική διαδικασία. Αυτό θα είναι σημαντικό πρόβλημα δεδομένου ότι η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες ε, στο μέλλον. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει δυνατότητα για τις μειονότητες να συμμετάσχουν και αυτές στη κυβέρνηση. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση να κάνει κάτι για να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις αυτές. Είχατε εις βάθος συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό σχετικά με το πώς σκοπεύει να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις πάνω στα ε, ανοιχτά κεφάλαια και θα ήταν δυνατά όλα αυτά με την μικρή πλειοψηφία που έχουν τώρα στο Κοινοβούλιο. Και μία ακόμη ερώτηση σχετικά με την ε, θρησκεία. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ε, μια συγκεκριμένη προσέγγιση στο θέμα αυτό. Ε, ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε από τη νέα κυβέρνηση. Θα είναι διατεθειμένη να καταργήσει το νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης. Και πιστεύετε ότι θα επιβραδύνει τη διαδικασία, ε, θα επιβραδύνει τη διαδικασία οι πολιτικές αντιθέσεις ε, που υπάρχουν. Αναφερθήκατε σε, στις επενδύσεις από τρίτες χώρες, ε, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς. Ε, κινδυνεύουμε εμείς να τεθούμε στο περιθώριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μάσιμο. Με ενημερώνουν ότι έχει συνδεθεί, τώρα ο Χέρμαν Τέρτς. Παρακαλώ, Χέρμαν. Γεια σας, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω σπανικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για την ενημέρωση. Είμαστε, δηλώνουμε, ικανοποιημένοι με τις εκλογές έτσι όπως διοργανώθηκαν στο Μαυροβούνιο. Ήταν ομαλές. Έχουμε μια πολιτική αλλαγή να δούμε πού θα οδηγήσει. Αυτό που πράγματι μας ανησυχεί είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας που θα είναι δραματική πάρα πάρα πολύ σύντομα. Διότι υπάρχει μια σειρά από χώρε που οπωσδήποτε επιθυμούν να παρέμβουν στα εσωτερικά πράγματα του Μαυροβουνίου και γνωρίζουμε πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στα Δυτικά Βαλκάνια. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν ποια μέτρα θα αναλάβουμε ώστε να υπάρξει ταχεία βοήθεια προς τη χώρα ώστε να αντιμετωπίσουμε ή να προλάβουμε αυτές τις εξωτερικές παρεμβάσεις από Κίνα, από Ρωσία, από Τουρκία, από όπου και να προέλθουν, να μην είναι τόσο βαριές, να μην είναι τόσο σοβαρές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τέατς. Τώρα ο εισηγητής, ο κύριος Πίτσουλα για το Μαυροβούνιο θα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ντέιβιντ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο που είναι σήμερα μαζί μας. Έχουμε πολύ κακή σύνδεση δυστυχώς. Αυτό που είναι μοναδικό σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μια νέα κυβέρνηση που θα διαμορφωθεί, έχουμε ένα σεβασμό των πολιτικών θεσμών και του κράτους δικαίου υπό αυτήν την έννοια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα πρέπει να βρει ένα modus operandi για να συνεργαστεί με τους ε, συνομιλητές μας. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας ε, με τις ε, δυνάμεις της αντιπολίτευσης και θα συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση, αλλά έχουμε μεγάλες προσδοκίες, ακόμα μεγαλύτερες, καθότι το 70 περίπου του εκλογικού σώματος υποστηρίζει την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρατηρήσαμε και μια ισχυρή διάσταση της συμμετοχής της Εκκλησίας, ακόμα και στο σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, και είδαμε και κάποιες επιθέσεις κατά μειονοτήτων μουσουλμανικής και άλλων σε γειτονικέ χώρες. Δεν ξέρω πώς τα εκτιμάτε όλα αυτά. Ως προς το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, δεδομένου του ότι έχουμε 7 από 7 εκπληρωμένες προτεραιότητες σχετικά με την πρόοδο της χώρας αυτής. Ελπίζω να σχηματίσουμε μία πλατφόρμα ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την πρόοδο της η χώρα. Η ερώτησή μου είναι τι προβλέπει η Επιτροπή σχετικά με τη νέα μεθοδολογία για τη διεύρυνση. Πώς αυτό θα έχει αντίκτυπο επί των διαπραγματεύσεων προσχώρησης. Η νέα κυβέρνηση έχει διαβιβάσει οποιοδήποτε σινιάλο για το πώς θα συνεχίσει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και ελπίζω να κλείσω πιο θετικά, πέρυσι είχατε πει όταν αναλάβετε τα καθήκοντά σας ότι ο στόχος σας ήταν μέχρι το τέλος της ε, εντολής σας, δηλαδή μέχρι το 2024, το Μαυροβούνιο να είναι έτοιμο να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι αυτό είναι ρεαλιστικός στόχος. Ευχαριστούμε τον κύριο Πίτσουλα. Συνάδελφοι, Έχουμε περιορισμένο χρόνο για το θέμα αυτό και το επόμενο θέμα είναι να ξεκινήσει 6 παρατέταρτο. Επομένως, λέω να μην ακούσουμε άλλους ομιλητές αυτή τη στιγμή, να ακούσουμε τον Επίτροπο, γιατί δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε και δεύτερο γύρο. Ε, παρακαλώ, δεχτείτε τη συγνώμη μου σχετικά με αυτό και Όλιβερ αν μπορείτε να μας απαντήσετε όσο πιο συνοπτικά γίνεται σε αυτές τις ερωτήσεις που έγιναν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ελπίζω να με ακούτε καλά. Να πάω πολύ γρήγορα στα ερωτήματα που ακούστηκαν ένα προς ένα. Σύμφωνο με τον κύριο Μπίλσικ ότι οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά. Και αυτό ήταν μια καλή βάση για την ανάληψη των καθηκόντων οποιασδήποτε νέας κυβέρνησης, αλλά και της πολιτικής αλλαγής στη χώρα. Η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση είναι πράγματι δεινή. Εμείς κινητοποίησαμε ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας και μακροοικονομική βοήθεια και δημοσιονομική συζητούμε, συνομιλούμε με διεθνείς οικονομικούς φορείς για περαιτέρω ενίσχυση εφόσον αυτή χρειαστεί, αλλά χρειαζόμαστε μια εκτίμηση και από πλευρά τη νέα κυβέρνηση σχετικά με το πώ ακριβώ έχει αυτή η οικονομική κατάσταση χώρας. χώρα. Θα καθίσουμε λοιπόν μαζί του να δούμε ακριβώ πώ έχει η κατάσταση, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε στη διάθεσή μα είναι μόνο εκτιμήσει. Τώρα για την καταπολέμηση του ιού αναμένοντας και το εμβόλιο που είναι σημαντικό χώρα για όλους μας θα είναι μέρος το Μαυροβούνιο ενός σχεδίου προμηθείας και θα έχουμε και δωρητές που στο προηγούμενο τρίμηνο είχαμε συμφωνήσει με αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και διερευνούμε πρόσθετες δυνατότητες εξασφάλισης επαρκούς αριθμού εμβολίων. Όταν θα έχουν τακτοποιηθεί όλες οι οικονομικές λεπτομέρειες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που το εξετάζουμε και το προετοιμάζουμε. Τώρα για πρόσθετα μέτρα προς τη βοήθεια που ρωτάτε. Σας επαναλαμβάνω ότι αυτή η εργασία τρέχει ακόμα. Θα πρέπει να συνομιλήσουμε και με τη νέα κυβέρνηση για το κατά πόσο επιθυμούν πρόσθετη ενίσχυση και τι μορφή θα είναι αυτή. Τώρα, πολλοί από εσά αναφερθήκατε στην έλλειψη μειονοτήτων στη νέα κυβέρνηση. Πράγματι, ισχύει και το έχουμε παρατηρήσει και παρατηρούμε και πολύ στενά την όλη κατάσταση στη χώρα διότι θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση και τη χώρα. Βέβαια δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε τι πλειοψηφία σχηματίζεται σε κάθε κοινοβούλιο και πώς σχηματίζεται. Υπογραμμίζουμε βεβαίως με τους συνομιλητές μας ότι είχε προστιθέμενη αξία εκπροσώπηση των μειονοτήτων προηγουμένως, μέχρι τώρα δηλαδή. Τώρα πώς μπορούμε να κλείσουμε κεφάλαια και να επιταχύνουμε την διαδικασία προσχώρησης. Αυτό εξαρτάται βεβαίως πάνω απ' όλα από την ίδια τη χώρα. Έχουμε πει με σαφήνεια ποιες είναι οι προτεραιότητες υπό τις οποίες θα μπορούσε να επιταχυνθεί η διαδικασία και ποια κεφάλαια θα μπορούσαν ακόμα να κλείσουν και βεβαίω το κεφάλαιο 23-24 του κράτου δικαίου είναι κλειδί. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε άλλα. Και θα πρέπει βεβαίω να δούμε και τα άλλα τεχνικά κεφάλαια για να πείσουμε τα κράτη-μέλη. Από πλευράς μας είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα Βεβαίως όλα εξαρτώνται, παραλαμβάνω, και από την συνεργασία με την κυβέρνηση της χώρας. Και επ' αυτού αναμένομαι. Τώρα, πώς έχουν οι με τη Σερβία. Η ένταση που είδαμε πριν από τις εκλογές έχει μειωθεί κάπως και ελπίζω να μειωθεί περαιτέρω, είναι αθετικό σημάδι ότι οι χώρες της γειτονία και η Σερβία και το Μαυροβούνιο παρακολουθούν αυτή την πρωτοβουλία της τοπικής κοινή αγοράς, το οποίο καταφέρνει να απαλύνει τις, ε, τις εντάσεις και τις πιέσεις. Τώρα εγώ δεν θεωρώ ότι το Μαυροβούνιο έχει δικαίωμα βέτο, όπως αναφέρθηκε, αλλά στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, συνεργασίας αυτής, αλλά θα χρειαστεί περαιτέρω συνεργασία για να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία. Δεν έχουμε κάτι τελικό αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε συμφωνία. Ακόμα φέτος. Ακόμα φέτος. για την κυρία Μπίλντε και τον κινέζικο αυτοκινητόδρομο κτλ. Ε, ναι, εντάξει. Ε, ε, συμφωνώ μαζί σας ότι τα έργα αυτά βεβαίως και έχουν αντίκτυπο επί των δημοσιονομικών της χώρας και υπήρξε και σημαντικό θέμα και στην προεκλογική εκστρατεία και θα είναι θέμα και για τη νέα κυβέρνηση που σχηματίζεται και επομένως θα δούμε πώς θέλουν να προχωρήσουν από αυτού. Σημαντικό μέρος της ε, πλειοψηφίας συνδέονται με το έργο αυτό. Από πλευράς μας, ώστε να βοηθήσουμε την οικονομία του Μαυροβουνίου και της Λιμπής περιοχής, δίνουμε βοήθειες και κίνητρα για έργα αντίστοιχης κλίμακας, ώστε να μπορέσει η χώρα και οι υπόλοιπε χώρες περιοχής να ανακτήσουν, να ενισχύσουν και πάλι την οικονομία τους μετά την κρίση. Εξετάζουμε και το θέμα των επενδύσεων σε κέντρα ενέργειας και ζητούμε και την απόσυρση, τη σταδιακή απόσυρση του άνθρακα. Ζητούμε από τις χώρες αυτές να μείνουν σε πλαίσια καθαρής ενέργειας και τελικώς να απομακρυνθούν τελείως από τον άνθρακα. Να γίνουν ουδέτερες ως προς τον άνθρακα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η νέα κυβέρνηση θα πιστεί από τα επιχειρηματά μας με, επί τη βάση των πρώτων επαφών που είχαμε τον κύριο Κρύβο Κάπιτς, νομίζω ότι υπάρχει διάθεση από πλευρά τους και θα πρέπει να τους το εξηγήσουμε όταν ελάβουν τα καθήκοντά τους και πιο ανοιχτά. Τώρα, ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε διαφορετική συμμαχία πολιτική που προκύπτει τώρα είναι ακριβώς τα θρησκευτικά ζητήματα. Πρέπει να έχουμε ελευθερία θρησκείας, πίστης, ανεξιθρησκεία εν πάση περιπτώσει στη χώρα. Πρέπει να είναι απόλυτα ελεύθεροι οι πολίτες να ασκούν, να ακολουθούν την, την δική τους ε, θρησκεία, τη δική τους εκκλησία χωρίς καμία πίεση από την πολιτική εξουσία ή αλλού. Είναι ένα θέμα το οποίο θα τεθεί στα πλαίσια της νέας συμφωνίας που θα έχουμε με το Μαυροβούνιο. Έχω συναντηθεί με τον κύριο Κρυβοκάπιτς. Αμέσως μετά την εκκίνηση του σχεδίου του οικονομικού και των επενδύσεων είχα την ευκαιρία να μιλήσω, να συζητήσω μαζί του σε ένα δείπνο επί μακρόν και η συζήτηση αυτή μου επιβεβαίωσε ότι είναι δεσμευμένος προς την ευρωπαϊκή κατεύθυνση πορεία της χώρας και ως προς την ε, συμμαχία με τον ΝΑΤΟ, κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μας για την ασφάλεια της περιοχής. Επί τη βάση λοιπόν της ανταλλαγής αυτής που είχα, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή που να προδιαγράφεται ως προς τις βασικές κατευθύνσεις της χώρας. Τώρα λυπάμαι ότι ίσως να μην μπορέσω να να απαντήσω σε όλες τις λεπτομερείς ερωτήσεις του κυρίου Βάιτσεν γιατί μάλλον είναι καλύτερο ενημερωμένος από μένα. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς θα χειριστεί το θέμα της ε, διαδικασίας προσχώρησης, αυτό που είναι σαφές για μας είναι ότι πρέπει να έχει σημαντική θέση, πρέπει να υπάγεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, Δηλαδή, για να το πούμε διαφορετικά, πρέπει να το βλέπει η νέα κυβέρνηση ως οριζόντιο θέμα για οποιαδήποτε πολιτική επιμέρους Υπουργείου. Αυτό θα ήταν καλό σημάδι για μας και ο αναπληρωτής Πρωθυπουργό, αν το αναλάμβανε θα ήταν καλό σημάδι. Θα του έδινε ε, τη θέση που του αξίζει του θέματος. Η κυβέρνηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της αυτό το οριζόντιο θέμα κάθε φορά που θα υπάρχουν αποφάσεις που θα μπορούσαν να το επηρεάσουν. Ο ρόλος τώρα του Προέδρου ο πρόεδρος έχει να διαδραματίσει έναν ρόλο σταθεροποίησης και ομαλότητας. Είχατε ευκαιρία να συζητήσω μαζί του. Μου είπε με σαφήνεια ότι είναι παρόν για να βοηθήσει, να συνοδεύσει αυτήν τη διαδικασία προσχώρησης και σχηματισμού της νέας κυβέρνησης και ότι αυτός από πλευράς του θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να συνεχίσει η χώρα προς την κατεύθυνση που είχε προδιαγράψει. Ο κύριος Καστάλντο νομίζω ότι ήδη απήντησα για το θέμα των μειονοτήτων και για την ανεκθρησκεία. Τώρα πώς μπορούμε περισσότερο να βοηθήσουμε αυτή τη τελευταία ερώτηση που κάνατε. το καλύτερο για μας είναι να έχουμε ένα θετικό θεματολόγιο. Με τη νέα μεθοδολογία λοιπόν και το νέο σχέδιο επενδύσεων έχουμε τα μέσα της θέσή μας για να έχουμε, να σχηματίσουμε ένα θετικό θεματολόγιο και κρίνοντας από τα όσα άκουσα και από την Ποντγκόριτσα και από αλλού στην ευρύτερη περιοχή αυτό το θετικό θεματολόγιο μπορεί και θα λειτουργήσει θα δίδονται ισορροπημένα αν θέλετε κίνητρα προς όλους και αυτό για μας είναι το βασικότερο. για τις παρεμβάσεις της εξωτερικής άλλων και πώς θα μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η περιοχή είναι η πιο κοντινή προς εμάς ε, και θα, πολύ δύσκολο θα μπορούσα να φανταστώ ότι κάποιος άλλος πιο μακριά θα μπορούσε να επηρεάσει πιο αποτελεσματικά. Είμαστε ο βασικός εταίρος της χώρας, αλλά αυτό επίσης σημαίνει ότι πρέπει να επιβεβαιώνουμε τον σημαντικό ρόλό μας στα μάτια της χώρας. Και επομένως είναι πολύ σημαντικό οικονομικά και πολιτικά για την όλη περιοχή, εκτός από τη χώρα, να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Θα εξακολουθήσουμε λοιπόν να πιέζουμε για περισσότερα και καλύτερα παραδοτέα, για τον κύριο Πίτσουλα. Ότι η έβδομη προτεραιότητα είναι το θέμα της ε, προσχώρησης. Η έβδομη από 7. Για την νέα κυβέρνηση δηλαδή. Εμένα με βεβαίωσαν ότι είναι η πρώτη της προτεραιότητα ιδιαίτερη δεδομένη της κατάστασης χώρας μετά το COVID ή εντό του COVID δηλαδή. Και μόλις με ενημέρωσαν ότι μάλλον η πρώτη επίσημη επίσκεψη του νέου Πρωθυπουργού όταν αναλάβει τα καθήκοντά του θα είναι μάλλον στις Βρυξέλλες. Και αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίσης σημάδι για τα κράτη-μέλη. Το κατά πόσον η νέα μεθοδολογία διεύρυνσης θα συμπεριλαμβάνει το Μαυροβούνιο και πώς είναι ένα πλαίσιο που θα μας βοηθήσει να ομαδοποιήσουμε τα συνδεδεμένα θέματα και να διαπραγματευόμαστε για περισσότερα πράγματα από κοινού εφόσον έχουμε παραδοντέα, εφόσον έχουμε δηλαδή πρόοδο. ο εντολοδόχος Πρωθυπουργό με βεβαίωσε ότι είναι έτοιμοι να επιταχύνουν τις δικές τους εργασίες και η νέα μεθολογία πιστεύω ότι είναι το κατάλληλο πλαίσιο. Θα μείνω εδώ προς το παρόν. Thank you. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Και σας ευχαριστώ που σταματήσατε ακριβώς την ώρα που είχαμε πει. Έξι παρατέταρτο. Νομίζω, συνάδελφοι, ότι είχαμε ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για το Μαυροβούνιο. Δυστυχώ δεν μπορώ να δώσω το λόγο στου άλλους συναδέλφους, γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε τώρα. Είναι η ώρα να συζητήσουμε για τη Σερβία. Και 6.30 θα πρέπει να τελειώσει η συνεδρίαση. Και προχωρούμε στο θέμα υπαριθμών 11. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, Επίτροπε. Α συζητήσουμε τώρα την κατάσταση στη Σερβία Παρακολουθήσαμε όλοι τις εκλογές της 21 Ιουνίου. Εκλογές που έγιναν παρά την πανδημία ε, του κορονοϊού. Ήταν χαμηλότερη η προσέλευση των ψηφοφόρων και έδωσε ε, πολύ μεγάλη πλειοψηφία στον σημερινό κυβερνητικό συνασπισμό και προς μεγάλη μας λύπη πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τις εκλογές. Στο μεταξύ ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση με προτεραιότητα ε, μεταξύ άλλων την ένταξη. Ωστόσο θα είναι μικρότερη η θητεία της κυβέρνησης γιατί εξήγηλε προκήρυξε, μάλλον εξήγηλε νέες εκλογές ο πρόεδρος Βούτσης πριν το τέλος του 2022. Εμείς ε, διευκολύναμε το διάλογο, το διακομματικό και έχει αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις η σημερινή κυβέρνηση που προτίθεται να τις υλοποιήσει. Ελπίζουμε να εξακολουθούν οι σερβικές αρχές να δείχνουν επικοδομητική στάση και προσήλωση και να μπορέσουν να συμφωνήσουν διμερώς και με το ε, Κόσοβο όπως και με το Μαυροβούνιο θα κάνουμε και εμείς έκθεση και για τη Σερβία 2019-2020. Το σχέδιο έκθεσης ε, κυκλοφόρησε ε, σήμερα το απόγευμα από πλευράς μου. Σταματώ εδώ και δίνω το λόγο στον Επίτροπο για 10 λεπτά για να μας μιλήσετε για την κατάσταση στη Σερβία. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Επίτρεψτε μου να έρθω τώρα στη Σερβία. Όπως Είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση, τα Δυτικά Βαλκάνια είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την περασμένη εβδομάδα η Σύνοδος Κορυφής στη Σόφια ήταν άλλη μία απόδειξη ότι το μέλλον όλης της περιοχής ε, είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι στρατηγικό μας συμφέρον να φέρουμε την περιοχή εκεί εντός της Ένωσης το συντομότερο και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο να διαδραματίσει εκεί η Σερβία. Είναι ο σημαντικότερος εταίρος μας εμπορικός. 60-65% όλου του εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης. Είμαστε και ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της Σερβίας και ο μεγαλύτερος επενδυτής. Έχει μια σαφή προοπτική ένταξης. 16 κεφάλαια έχουν ανοίξει και δύο έχουν κλείσει προσωρινά στις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω όμως ότι η Σερβία φέρει μοναδική ευθύνη για να αποδείξει ότι συνεχίζει μπροστά στο, στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η νέα σερβική κυβέρνηση, με πρωθυπουργό την Άννα έχει πάρει μεγάλη ψήφο εμπιστοσύνη στη Σερβική Βουλή, αλλά και από το λαό το καλοκαίρι τη λαϊκή ετοιμιγορία. 24 μέλη έχει νέα κυβέρνηση, 11 γυναίκες και 3, 3 νέα υπουργεία έχουν δημιουργηθεί μεταξύ αυτών Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαλόγου με την Κοινωνία. Πολύ ενθαρρυντικό ότι η νέα κυβέρνηση θέλει να συνεχίσει το διάλογο με το Κόσοβο ε, ως δεύτερη προτεραιότητα και, πρώτη προτεραιότητα ε, ε, ε, είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά πολύ ψηλά επίσης η καταπολέμηση της πανδημίας. Ενδιαφέρουν αυτά πάρα πολύ το σερβικό λαό. Είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσει στο δρόμο αυτό η κυβέρνηση και όπως είπε και ο Πρόεδρος, και ε, η νέα Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση αυτή, είναι μια κυβέρνηση μεταρρυθμίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πλήρως προσιλωμένη στην υποστήριξη της Σερβίας σε αυτό το δρόμο. Δώσαμε και 15 εκατομμύρια για τις άμεσες ανάγκες της πανδημίας, για προμήθεια υλικού ε, ιατρικού εξοπλισμού, υποστήριξη ευάλωτων ατόμων στην κοινωνία και ομάδων και κατεξαίρεση πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού για να ε, ανακουφιστεί λίγο η πίεση. Προβλέπουμε και άλλες ε, δαπάνες για κάλυψη πρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών για την πανδημία, για την υποστήριξη οικονομικής ανάκαμψης τις δραστηριότητες ε, βοήθησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του τουρισμού που έχει πληγεί σφοδρά με ιδιαίτερη προσήλωση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Πιο μακροπρόθεσμα θα υποστηρίξουμε την ε, οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη και σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν έχει και καλύτερες συνδέσεις αεροπορικές και οδικές, ε, θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις ε, απασχόλησης για την κομβική η Σερβία στην περιοχή. Επίσης, στόχος είναι να αυξηθεί η ποιότητα ζωής του πληθυσμού στις πόλεις. Η ενίσχυση των επενδύσεων όμως και της οικονομικής ανάπτυξης στα Δυτικά Βαλκάνια θα γίνει μόνο εφόσον γίνουν οι βασικές θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις οικονομικές, ενίσχυση κράτους δικαίου, βελτίωση της δημοσίας διοίκησης. Είναι εκ των όνων κάνευ αυτές οι μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για τον ευρωπαϊκό δρόμο της Σερβίας, αλλά και για να δημιουργηθεί αξιόπιστο και βιώσιμο επενδυτικό κλίμα. Τον Οκτώβριο εγκρίναμε μια έκθεση που θα βρείτε εκτενή επισκόπηση της ε, ε, κατάστασης και των βημάτων που πρέπει να γίνουν παραμένει θεμελιώδες να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια με τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για την ενταξιακή πορεία, αλλά για να πετύχει και το σχέδιο για την οικονομία και τις επενδύσεις. Πρόσφατα μετέβαινε στη χώρα και ενθάρρυνα την κυβέρνηση να αξιοποιήσει όσο γίνεται καλύτερα την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομία, οικονομία και την ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι θετικές οι εξελίξεις. Πριν από την κρίση ε, ε, είχε μπει σε γερή οικονομική ανάπτυξη η Σερβία και βλέπουμε ότι είναι η χώρα όπου η πανδημία ε, του κορονοϊού έπληξε λιγότερο την οικονομία. Χάρη στο γενναίο όδωρο πακέτο στήριξης της κυβέρνησης αποσοβήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι αρνητικές συνέπειες. Βεβαίως, έχει μειωθεί η παραγωγικότητα και η απασχόληση, αλλά η χώρα τα βγάζει καλύτερα πέρα από ε, την υπόλοιπη περιοχή. Συνέχισε λοιπόν το μεταρρυθμίσεων με βιώσιμο τρόπο. Αυτό θα απαιτήσει ένα γνήσιο διάλογο σε όλο το πολιτικό φάσμα και με την ισχυρή εντολή της νέα εκλεγής σας ε, Βουλής ελπίζουμε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα η κυβέρνηση όλες τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να ε, προχωρήσει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω τη συνεχιζόμενη επικοδομητική στάση για την περιφερειακή συνεργασία είναι υψής της σημασίας. Το είδαμε και στη Σόφια την περασμένη εβδομάδα. Η κοινή περιφερειακή αγορά που εγκρίθηκε θα είναι πολύ σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή πορεία και της Σερβίας και της περιοχής. Θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα και θα ε, κάνει ελκυστικό προορισμό επενδύσεων τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτές και άλλες μεταρρυθμίσεις θα ανοίξουν το δρόμο και για νέα κεφάλαια, να ανοίξουν νέα κεφάλαια στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, κάτι το οποίο περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο για τη στήριξη και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Βαρχέλη. Σχετικά με την ενημέρωση, σχετικά με τη Σερβία από τη δική σας οπτική. Περνάμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων. Με ενημερώνουν ότι ο επικεφαλής της, η, επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, για τις σχέσεις με τη Σερβία, η Τάνια Φαγιών, δεν μπορεί να είναι παρούσα απόψε. Οπότε δίνω το λόγο ε, στον εκπρόσωπο του ΕΛΚ κατευθείαν. Παρακαλώ. elections will be held on April 3 Απριλίου του 2021 θα πραγματοποιηθούν εκλογές, ε, το οποίο σημαίνει ότι η, η ε, παρούσα κυβέρνηση έχει 1,5 χρόνο συνολικά θητεία. Ε, θέλουμε ωστόσο να διασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό μέλλον της Σερβίας και η Έχω την εξή ερώτηση. ω μέρο ε, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η ευθυγράμμιση της ε, κοινή ε, αμυντικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλή δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Η χώρα δεν είναι απόλυτα προετοιμασμένη για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Ε, κατά 60% ήταν προετοιμασμένοι το 2019 και φυσικά ο βασικός στόχος είναι η ειρήνη και η ασφάλεια. Πώς σκοπεύετε να εξηγήσετε στη Σερβία ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ε, να εργαστούμε όλοι για έναν για να μπορούμε να σεβαστούμε ε, τον, ε, την κοινή πολιτική ασφαλείας μας. Ευχαριστώ πολύ για την σύντομη αυτή παρέμβαση και δίνω το λόγο στον Τονίνο Πίτσουλα από το S&D. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Ντέιβιντ. Ε, κύριε Επίτροπε, κατευθείαν θα περάσω στο θέμα που με ενδιαφέρει. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τις ανησυχίες μας για την κατάσταση στη Σερβία. Ε, όσον αφορά τις νέες τάσεις, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην οπισθοχώρηση όσον αφορά ε, την δημοκρατική λογοδοσία, το κράτος δικαίου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, ε, καθώς και τον αυξανόμενο ευροσκεπτικισμό. Η έκθεση προόδου για την ε, Σερβία ε, εν μέρη αντικατοπτρίζει αυτή την έλλειψη ε, προόδου. Τονίνο, you are unfortunately... Το δυστυχώς κόπηκε η σύνδεση, δεν σε βλέπουμε, δεν σε ακούμε. Τώρα με βλέπετε. Ναι. Ωραία, θα προσπαθήσω να συντομεύσω. Δικαίω θα μπορούσε να πει κανεί ότι η αντιπολίτευση μποϊκοτάρισε τι εκλογέ και εμεί ω πολιτική ομάδα πάντα ενθαρρύνουμε όλου να ε, συμμετέχουν στι κοινοβουλευτικέ εργασίε. Ωστόσο, την προεκλογική περίοδο στην ε, Σερβία ε, η η κυβέρνηση δεν δέχτηκε γενέστερη ημερομηνία για τις εκλογές όπως, είχαν, όπως είχε προτείνει η σοσιαλιστική ε, αντιπολίτευση. Ενώ σε άλλη περίπτωση είχαμε δεχτεί μια τέτοια αναβολή που έγινε αποδεχτή από την κυβέρνηση. 29 συστάσεις ε, περιέχει η ε, έκθεση ε, για την Σερβία παραπάνω από για οποιαδήποτε άλλη χώρα την τελευταία δεκαετία. Δεν υπάρχει ουσιαστική αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο, από ό,τι γνωρίζω. Είναι η πρώτη περίπτωση χώρας υποψήφιας για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο τον ε, Ιούλιο 37 μη κυβερνητικέ οργανώσεις και 20 άτομα ε, τέθηκαν υπό έρευνα για πιθανό ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση ε, τρομοκρατίας. Κυρίως πρόκειται για οργανώσεις και δημοσιογράφους που είναι επικριτικοί απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Ε, θα πρέπει να ζητήσουμε τουλάχιστον εξηγήσει. Ε, κύριε Επίτροπε, έχετε ζητήσει κάτι τέτοιο, έχετε ζητήσει σχετικέ εξηγήσει. Σα ευχαριστώ προκαταβολικά για τι απαντήσει σα. Ευχαριστώ πολύ τον Νίνο. Ιλάν Κούτσουκ, παρακαλώ. Chair, thank you. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο απόψε. Παρουσιάσατε την ετήσια έκθεση για τη Σερβία μαζί με το επενδυτικό σχέδιο. Η γενική αξιολόγηση είναι ότι η Σερβία προοδεύει όσον αφορά την οικονομία, όχι όμως όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει έλλειψη προόδου όσον αφορά ε, τον δικαστικό τομέα, την ελευθερία μέσων ε, μαζικής ενημέρωσης, την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, κλπ. Επίσης είχατε αναφέρει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ανοίξει ε, το κεφάλαιο 8 για την πολιτική ανταγωνισμού. Έχοντας κατά νου όμως ε, τις ε, συστάσεις της έκθεσης, τι πιθανότητες υπάρχουν να ανοίξει νέο κεφάλαιο η Σερβία, ιδιαίτερα εφόσον ο πρόεδρος Βούλσης έχει τη συγκεκριμένη στάση που έχει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θέση που κράτησε κατά τη διάρκεια της κράσης του κορονοϊού τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από το ID Thierry Μαριάννη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Okay, Monsieur Mariani is not connected. Δεν ε, έχει συνδεθεί ο κύριος Μαριανή. Προβλέπεται αντικαταστάτρια που είναι η κυρία Ζουλή Chanteux. Είστε στη σύνδεση. Κυρία Λουσόντου, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ο σερβικός λαός είναι ιστορικός φίλος της Γαλλίας και ανέκαθεν ε, ε, κρατούσε το λόγο του και στο πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν στο πλευρό μας. Θέλω να επανέλθω στο διάλογο ε, βελιγράδι, πριστινα που ε, υποτίθεται ότι θα λύσει τις διαφορές ε, Σερβίας και της λεγόμενου Κωσόβου. Είναι σερβική επαρχία, Κόσοβο μετόχια, Κωσυφοπαίδιο ε, και είναι και ε, προϋπόθεση το έχετε βάλει για να μπει στην Ένωση η Σερβία. Με ποιο δικαίωμα. Πώς μπορείτε να ζητήσετε από τη Σερβία να αναγνωρίσει το Κόσοβο όταν υπάρχουν ακόμα πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανία, Ρουμανία, ε, Κύπρος, Ελλάδα και Σλοβακία που δεν το αναγνωρίζουν και καλά κάνουν γιατί ε, ο υποτιθέμενος πρόεδρος ε, ε, προσωρινά κρατείται εν ώψη δίκης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σας ευχαριστώ. Merci, Madame Ευχαριστώ κύριε Λεσόντε. Και τώρα από τους Πρασίνους η Βιόλα Φον Κράμον Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Έχω κάποιες ερωτήσεις για την υποχώρηση της δημοκρατίας στη Σερβία. Θα βάλετε νέα ορολογία στην έκθεση προόδου. Δεν είναι απλώς όχι, η έλλειψη προόδου. Είναι υποχώρηση της δημοκρατίας και επειδή υπάρχει και μια νέα μεθοδολογία, βλέπετε τίποτα εκεί. Η στρατηγική για τη διεύρυνση έχει και κάποιες εξωτερικές ε, παραμέτρους. Υπάρχουν ε, ορισμένοι που θέλουν να κρατηθούν στην εξουσία. Και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δέχεται κάποια σχετικοποίηση ε, ε, και ολίσθηση που φέρνει τη Σερβία πιο κοντά σε μια αυταρχική αντιδημοκρατική κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δει υποψήφιες χώρες να αναπτύσσουν ε, δημοκρατικές κυβερνήσεις. Πώς θα αντιστραφεί αυτή η αρνητική τάση που διαφαίνεται στη Σερβία. Και θέλω να ρωτήσω κάτι για τους Αλβανούς στο νότο αλβανικής καταγωγής Σέρβου, στο νότο της Σερβίας, ε, περίπου 4.000 έχουν αφαιρεθεί από το δημοτολόγιο. Ε, τι, θα κάνετε εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Thank you, Viola. Ευχαριστώ, Βιόλα. Ο κύριος Τέρτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με αυτήν την οπισθοδρόμηση που αναφέρουμε αυτές τις ανησυχίες δηλαδή για των τεκτενομένων στην Σερβία για, την, για τις οποίες όλοι μιλούν λέει ο μιλητής εσείς έχετε δει στις επαφές σας κάποια θετική ανταπόκριση σε αυτές τις ανησυχίες που εκφράζουμε εμείς εδώ που και που και εσείς εκφράσατε. Επίσης μπορείτε να μας πείτε ποια ήταν η αντίδραση του Βελιγραδίου στις έντονες ανησυχίες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά που περνούν πάντοτε μέσα από το Βελιγράδι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, τον κύριο Τέρτς, για, το... για την ΚΟΕ. Εμμανουέλ Μορέλ είναι συνδεμένος. Παρακαλώ. Κυρία Μορέλ, θα κάνουμε ένα refresh στη σελίδα σας, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Κύριε Μορέλ, δεν σας ακούμε, λέει ο πρόεδρος. On pas Προσπαθεί ο πρόεδρος να πει στα γαλλικά, δεν σας ακούμε. Okay, Monsieur Morel, um, on ne peut pas entendre. Νέα προσπάθεια του Προέδρου να πει στα γαλλικά στον κύριο Μορέλ ότι δεν τον ακούμε. Α πάω στον επόμενο μιλητή, στου μη εγγεγραμμένου, ο κύριο Καστάλλο. Ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ Πρόεδρε και τον Επίτροπο Βαρχελή για την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή του για ένα θέμα που είναι σημαντικότατο για την Ένωσή μας. Η ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό όραμα δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι ότου να προσχωρήσουν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Υπάρχουν ιστορικοί και παραδοσιακοί λόγοι που εξηγούν κάτι τέτοιο και υπάρχει και σημαντικό διεθνές διακύβευμα. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν κάποια εμπόδια και η σερβική περίπτωση είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρά τις θετικές εξέλιξεις των τελευταίων ετών, το Βελιγράδι θα πρέπει να υιοθετήσει ένα θεματολόγιο φιλόδοξο ε, προσχώρησης μαζί με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει προς την κατεύθυνση αυτή και εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ε, εκτός από τις εξωτερικές πιέσεις και επιρροή που έχουμε και που πρέπει να δούμε. Και θα ήθελα να ρωτήσω τα εξή δύο ως προς αυτό. Με την κρίση του COVID είδαμε στις διμερείς σχέσεις ε, μια ιντεντικοποίηση μεταξύ Βελιγραδίου και Πεκίνου το οποίο κατέληξε σε μια ρητορική σε τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων και άλλων στα μέσα ενημέρωση Σερβία με έναν τρόπο φιλοκινέζικο και αντιευρωπαϊκό, με συγχωρείτε, μήπως αυτό ζημιώνει τις ε, προσδοκίες της χώρας προς την ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Επίσης, οι σχέσεις μας με την Σερβία και το Κόσοβο φαίνεται να βασίζονται σε μια αμφιλεγόμενη συμφωνία που έγινε με την κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα, μαζί με τους εκπροσώπους από το Θάτσι, μάλλον του κυρίου Θάτσι. Ποια στάση μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες και τι μπορούμε να περιμένουμε από την διακυβέρνηση Biden στα πλαίσια αυτής της, ε, του μέλλοντος αυτής της διαπραγματεύσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Φάμπιο. Ο μόνιμος ηγητής μας, ο κύριος Μπίλτσικ, έχει τώρα το λόγο. very uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, David. Ευχαριστούμε για την Επίτροπο για την εισήγησή του. Συζητούμε σήμερα δύο χώρες που ηγούνται στην όλη περιοχή και σε περιοχές πολιτικής που είναι προς το στρατηγικό μας ε, συμφέρον. Μιλούμε πράγματι για θέματα διεύρυνσης και προσχώρησης και με το ίδιο επικοδομητικό με συγχωρείτε πνεύμα που μίλησα και για το Μοβροβούνιο θέλω να μιλήσω και για τη Σερβία. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Νομίζω ότι έχει διανυμηθεί και στα μέλη της Επιτροπής το σχέδιο της νομοδότησής μου και στα πολλά ερωτήματα και παρατηρήσεις που ήδη αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους θα ήθελα να προσθέσω ότι περιμένω μεγάλο ενδιαφέρον για τις πολλές και δύσκολες συζητήσεις πρέπει να έχουμε για το μέλλον της Σερβίας, διότι, ε, ξαναλέω, εδώ συζητούμε για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, συζητούμε για τη διεύρυνση. Αυτό είναι ο τρόπος να συνομιλούμε και με τη νέα κυβέρνηση της Σερβίας, την οποία χαιρετίζουμε, και τη νέα σύνθεση της Βουλής, που σχηματίστηκε υπό δύσκολες συνθήκες, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί προς την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Περιμένουμε ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει τις εποχές της και θα τις τηρήσει αποφασιστικά. Ρωτώ λοιπόν Επίτροπε, η δική σας εκτίμηση των συζητήσεων στο Συμβούλιο ποια είναι. Το Συμβούλιο είναι έτοιμο να ανοίξει και άλλα κεφάλαια για τη Σερβία. εφόσον η Σερβία τηρήσει αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. Και απαντώντας σε κάποια σημεία που έθιξαν οι συνάδελφοι για το διακομματικό διάλογο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι δεσμευμένο προς διακομματική συζήτηση και διάλογο, ο οποίος έχει επιφέρει και πολύ απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μαζί με τους συναδέλφους νομίζω ότι έχουμε επιτύχει Δεσμεύσει από πλευρά των ε, Σέρβων. Έχουμε επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, συγκεκριμένη πρόοδο ακόμα και στο πλαίσιο των εκλογών. Αυτό πρέπει να το εξακολουθούμε να το κάνουμε και για τις ε, μελλοντικές εκλογές το 22 και αυτό πρέπει να το κάνουμε επικοδομητικά. Να υπερασπιζόμαστε δηλαδή τις ευρωπαϊκές μας αξίες και αρχές, τα κριτήρια για τη διεύρυνση και να συνεχίζουμε το διάλογο με τους εταίρους μας. Πολύ λυπούμε ότι ένα μέρος αντιπολίτευσης δεν συμμετείχε σε εκλογές αυτές. Ελπίζω να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περιοχή για αυτές στο μέλλον. ώστε να έχουμε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές με συνολική συμμετοχή όλων και υπολογίζουμε και στην ελπίδα του Επιτρόπου για να διευκολύνει το διάλογό μας με τους ε, Σέρβους πολιτικούς και στην προσπάθειά μας να εξωθήσουμε για μεταρρυθμίσεις, αλλαγές, το, την ευρωπαϊκή προοπτική και μέλλον της χώρας. Χρειαζόμαστε θετικά σημεία και από το Πελιγράδι αλλά και από το Συμβούλιο. ώστε αυτές οι θετικές αλλαγές να λάβουν χώρα Σερβία όσο δύσκολο και να φαίνεται κάποιες στιγμές περιμένουμε με ενδιαφέρον συνέχιση τη ζήτηση για το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ, Βλάντιμιρ. Θα, προσπαθούμε, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον Εμμανουέλ Μορέλ. Παρακαλώ. Κύριε Μορέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Σας ακούμε, αλλά έχει πολύ αέρα. Δεν θα μακρηγορήσω για την πολιτική κατάσταση στη Σερβία, γιατί οι συνάδελφοι ε, αναφέρθηκαν σε εκλογές αυτές και την αποχή της αντιπολίτευσης, που είναι λυπηρό γιατί ακόμα και αν ήταν κανονικές οι εκλογές, είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ένα κοινοβούλιο που δεν εκπροσωπεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεισφέρει στο να εδραιώσει ένα διάλογο ανάμεσα στο κόμμα του Προέδρου Βούτσιτς και την αντιπολίτευση. Θέλω να αναφέρω κάτι που δεν ακούστηκε μέχρι τώρα. Συχνά ε, συζητούμε για τις σχέσεις Σερβίας-Ρωσίας, που είναι ιστορικές, πολιτισμικές και κανονικές, θα έλεγα, φυσιολογικές. Από την άλλη όμως θέλω να μιλήσουμε για την Κίνα, γιατί υπάρχει μια κινέζικη στρατηγική στην ε, Σερβία που θα πρέπει να μας ανησυχεί. Ε, είναι στο στόχαστρο της Κίνας η Σερβία. Τη θεωρεί σημαντικό άξονα για το νέο δρόμο του μεταξιού και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει ρόλο εκεί γιατί μας ενδιαφέρει η γειτονία μας και η όλη επικοινωνία ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης της Κίνας. Ξέρουμε ποια είναι, έστειλαν ιατρικό υλικό, πολύ καλά πήγε. Στην Ευρώπη όχι, στην αρχή ε, μπλοκαρίστηκαν και όλες από τις Βρυξέλλες οι εξαγωγές υλικού. Τελικά της δόθηκε βοήθεια, αλλά ε, πολλές εβδομάδες ε, μετά την προσγείωση κινέζικων αεροπλάνων κάργο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει τη Σερβία ότι είναι σημαντικός εταίρος, αξιόπιστος εταίρος και μόνο έτσι η Σερβία θα ανακτήσει πλήρως την ευρωπαϊκή της ε, ε, μοίρα, τουλάχιστον εμείς αυτό επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, όπως και προηγουμένως για το Μαυροβούνιο, έχουμε καθυστερήσει, δεν θα δώσω το λόγο σε άλλους συναδέλφους. Ακούσαμε ένα γύρο των ε, συντονιστών και το μόνιμο εισηγητή. Θα δώσω το λόγο πάλι στον Επίτροπο για να τελειώσουμε σε 10-12 λεπτά. Αν μπορείς για 10 λεπτά, Όλιβερ, ε, ε, να συνοψίσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Ντέιβιντ. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις απαντήσεις ε, για να είμαι κάπως σύντομος. Καταρχάς, όσον αφορά τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση και την προσήλωσή της στις μεταρρυθμίσεις. Πώς βλέπουμε το θέμα. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η κυβέρνηση σχηματίστηκε σύμφωνα με τη δική μας ερμηνεία και Αυτά κατάλαβα από τη συνάντηση ε, με τον κύριο Βούλση αλλά και με τον Πρωθυπουργό ότι η ε, κυβέρνηση αυτή είναι κυβέρνηση μεταρρυθμίσεων που στόχο έχει να εφαρμόσει τις ε, μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό τώρα εξετάζουμε έναν κοινό οδικό χάρτη για να επιταχύνουμε τις εργασίες. Νομίζω ότι η προσήλωση είναι απόλυτη από τη δική τους πλευρά. Αύριο θα συναντηθώ με τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που νομίζω θα μου περιγράψει και τα σχέδιά τους. Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν έχει την απαραίτητη κοινοβουλευτική υποστήριξη και εξουσία για να παρουσιάσει αποτελέσματα. Είναι μοναδική η ευκαιρία αυτή, την οποία θα πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε, όχι μόνο για τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί και μοναδική ευκαιρία για να έχουμε τον διάλογο ε, Βελιγραδίου και Πρίστινας ε, και να επιτύχει ο διάλογος αυτός. Ε, θα καλώ λοιπόν όλους που μπορούν να συνεισφέρουν να το κάνουν αυτό και να εκμεταλλευτούν στο έπακρον ε, τα δύο αυτά χρόνια που έχουμε στη διάθεσή μας, διότι πιθανότατα να μην ξαναέχουμε μια τέτοια ευκαιρία στο εγγύς Όσον αφορά την οπισθοδρόμηση και τις επικρίσεις, πράγματι Είχαμε μία ε, περίοδο με ε, πολύ αργές εξελίξεις, ε, ωστόσο η κυβέρνηση συνέχισε να εργάζεται πάνω σε τομείς όπου μπορούσε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις δεδομένου ότι είχαμε και τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Ο σχηματισμός της κυβέρνησης ε, απέτησε περισσότερο χρόνο από το περιμέναμε. Τώρα όμως υπάρχει δυνατότητα να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις. Η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα είναι υψίστης σημασίας. Υπάρχει τώρα πια πλειοψηφία υπέρ της κυβέρνησης. Ελπίζω λοιπόν η κυβέρνηση σύντομα να μπορεί να παρουσιάσει αποτελέσματα. Επίσης ε, βλέπουμε ότι πρέπει να γίνουν πράγματα όσον αφορά την ε, ανεξαρτησία των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με χαρά μπορώ να σας ενημερώσω ότι η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει εργασίες πάνω στη νέα στρατηγική για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία θα εφαρμοστεί και με τη δική μας οικονομική υποστήριξη. Περιμένω να δοθεί θετική ορμή με όλα αυτά. Ναι, έχουμε τις ε, συστάσεις ε, του ΟΑΣΕ, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι τις επόμενες εκλογές. Είμαι αισιόδοξο ότι η διετία αυτή θα είναι μια διετία ε, σκληρής εργασίας και καλών αποτελεσμάτων και έτσι φτάνω στην επόμενη ερώτηση. Έτσι θα μπορέσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη μας να ανοίξουν όλα τα απαραίτητα κεφάλαια για πιο ταχεία διαδικασία προσχώρησης, αλλά και για να αρχίσουμε να κλείνουμε κεφάλαια με τη χώρα. Όπως είπα, έχουμε μοναδική ευκαιρία μπροστά μας και νομίζω ότι το γνωρίζει αυτό και η κυβέρνηση. Η δεύτερη μεγάλη ομάδα θεμάτων σχετιζόταν με τις ε, εξωτερικές επιρροές και το πόσο ευάλωτη είναι η χώρα. Απέναντι σε αυτές είναι μια παρατήρηση που ακούω συνέχεια. Από το Μάρτιο ακούω ε, παρατηρήσεις ε, σχετικές ε, με ε, τον κορονοϊό και τον πρόεδρο οι συνάδελφοι που τα επαναλαμβάνουν όλα αυτά ε, αγνοούν τις κοινέ προσπάθειες και την κοινή μας επένδυση και ξεχνάνε, παραβλέπουν ότι ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση μας ευχαριστούν, συνεχίζουν να μας ευχαριστούν για όλα όσα κάναμε. Διότι εμείς παρήχαμε το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας τελευταία φορά που με ευχαρίστησαν δημοσίως ε, ήταν κατά την επίσκεψή μου τον Οκτώβριο στο Βελιγράδι. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι καλή ιδέα να ε, παρατονίζουμε το θέμα αυτό. Η, βοήθεια είναι βοήθεια, δεν είναι ε, αγώνας δρόμου. Δεν είναι ανταγωνισμός. Παίζουμε λοιπόν θετικό ρόλο, όχι μόνο ε, στα μάτια των κυβερνώντων ε, στη Σερβία, αλλά και γενικότερα. Για μένα λοιπόν θα συνεχίσει αυτό να είναι ένα καλό παράδειγμα, ε, κάτι θετικό από όλη αυτή την κρίση του κορονοϊού. Και κάτι πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε την εφαρμογή του οικονομικού και επενδυτικού προγράμματος. Τα επόμενα τέσσερα με πέντε χρόνια θα πρέπει να πείσουμε τους ε, ανθρώπους της Σερβίας ότι εμείς είμαστε ο πιο σημαντικός εταίρος, ότι εμείς έχουμε την καλύτερη... Ε, εμείς μπορούμε να προσφέρουμε τα καλύτερα στην περιφέρεια αυτή και μπορούμε να συμβάλλουμε όχι μόνο στη γενική εικόνα, αλλά και στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Αυτήν βάζουμε στο επίκεντρο. δηλαδή ε, αποσυμφόρηση στα πιο βασικά προβλήματα, ε, σιδηροδρομικές και οδικές ε, συνδέσεις, διαδικτυακές συνδέσεις, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, πράσινη ενέργεια, μείωση των υψηλών χειμερινών εκπομπών που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες μέσω των ε, οποίων θα έχουμε και ήδη έχουμε ε, ένα θετικό αφήγημα. Γι' αυτό ανέφερα την ε, προστιθέμενη αξία της συνάντησης στην Σόφια και τη σημασία της ε, κοινή οικονομικής ε, ε, περιοχής που, δημιουργεί, που δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είμαστε στο πλευρό των Σέρβων και έτσι θα έχουμε θετική ορμή και όσον αφορά τη δική μας παρουσία εκεί. Όσον αφορά τον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε το σημαντικό ρόλο αυτόν. Στην Ουάσιγκτον, η, συνάντηση, η συμφωνία που επιτεύχθη ήταν ένα πρώτο βήμα και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές από τις ε, πρωτοβουλίες που προωθούμε αντικατοπτρίζονται και αυτές στη συμφωνία. Προωθούμε σημαντικές ε, οικονομικές ε, και σχέσεις και υποδομές και η ιδέα του οικονομικού χώρου στην περιφέρεια αυτή είναι κάτι που έχουμε προωθήσει. Βλέπω λοιπόν να μπορούμε να παίξουμε πολύ θετικό ρόλο και σε συνεργασία με τους φίλους μας στις Ηνωμένε Πολιτείε. Δύο χρόνια διαρκεί αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που μας παρουσιάζεται και είμαι πεπισμένος ότι μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείε θα το πετύχουμε αυτό. Χωρίς τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι σχεδόν αδύνατο να το πετύχουμε. Η δική μας αξιολόγηση λοιπόν είναι ότι έχουμε μια μοναδική ευκαιρία μπροστά μας και ας την εκμεταλλευτούμε στο έπακρον. Όσον αφορά τον διακομματικό διάλογο, πράγματι έχει σημαντικά ωφέλη και πιστεύω ότι το νέο κοινοβούλιο ε, θα είναι και αυτό προσιλωμένο στους ίδιους στόχους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Βέλτ και την κυρία Τάνια Φαγιόν για όσα έχουν πετύχει και λυπάμαι για το, μποϊκοτ, για το μποϊκοτάζ, διότι αυτό δεν είναι προς όφελος της σερβικής δημοκρατίας. αλλά αυτό το κοινοβούλιο έχουμε με το οποίο πρέπει να συνεργαστούμε και ελπίζω σε, δύο χρόνια να έχουμε πλήρη συμμετοχή όλων των πολιτικών εταίρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Συνάδελφοι. Υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να πάρει το λόγο. Πολύ λυπάμαι που είχαμε μόνο δύο γύρους συζήτησης 45 λεπτών ε, για τις δύο αυτές χώρες. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τον Επίτροπο που συμμετείχε στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Η ΑΦΕΤ θα συνεχίσει τις εργασίες πάνω στην έκθεση για τη Σερβία 2019-2020. Το σχέδιο έκθεσης θα εξεταστεί στις 10 Δεκεμβρίου. 15 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ 4 Φεβρουαρίου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Μάρτιο. Οι επόμενες μας συνεδριές θα πραγματοποιηθούν 2 Δεκεμβρίου από τις 2 και 4 με 4 και 4 και από 5 και 4 με 7 και 4 και στις 3 Δεκεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 12 και από τις 2 παρατέταρτο μέχρι τις 4 παρατέταρτο και από τις 5 παρατέταρτο μέχρι τις 7 παρατέταρτο. Και πάλι αυτό οφείλεται στα, στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας λόγω του κορονοϊού. Αυτά από μένα. Κλείνω τη σημερινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους ε, για τη συμμετοχή τους.